Ja, meine lieben Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας αυτό το απόγευμα. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Από από, από το αρχικό στάδιο στην έναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους σήμερα ανάμεσά μας και θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω τον ε, κύριο Τιμ Γκρόσερ, Υπουργό Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, τον Justin Brown, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για εμπορικά ζητήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας. τον κύριο Μαρκ Χίγκη από την Αυστραλία, πρέσβευτη στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και τον David Τέιλορ, πρέσβη της Νέας Ζηλανδίας. Επίσης έχουμε μαζί μας τον κύριο Πασκάλ Κέσνάης, διευθυντή του European Services Forum, τον κύριο Μακιγιάμα, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, τον κύριο Πέκα Πέσονεν, Γενικό Γραμματέα της ΚΟΠΑ. Καλώς ήλθατε λοιπόν όλοι. Γνωρίζετε ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν ιδιαίτερα στενές εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστραλία συμμετέχει στην συμφωνία TPP και η Αυστραλία με τη Νέα Ζηλανδία διεξάγουν συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που είναι και η αφορμή και η βάση της ε, σημερινής μας συζήτησης. Και θα ήθελα, λοιπόν, να δώσω το λόγο τώρα στους ε, δύο πρέσβεις, ο καθένας για πέντε λεπτά, έτσι ώστε να μας κάνουν τα εισαγωγικά του σχόλια για το πάνελ που έχουμε σήμερα. Κύριε Χίγκη, έχετε πρώτο το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, να συμμετέχω σε αυτήν την δημόσια ακρόαση. Ε, με χαρά μου βλέπω γνώριμα πρόσωπα από την ομάδα παρακολούθηση Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, καθώς και ε, μέλη της αποστολής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθώς και τους συναδέλφου, μου, κύριο Γκρέσο και Τέιλορ. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κύριος Μπράουν θα κάνει στη συνέχεια ορισμένα ε, σχόλια και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που θα πει ο Τζάστιν με κάποια γενικότερα σχόλια για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Πριν από δύο εβδομάδες έλαβε χώρα η πρώτη σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας τα τελευταία ε, πέντε χρόνια. Συζητήσαμε στα πλαίσια της ε, συνόδου G20 στην Τουρκία συζητήθηκαν τα στάδια πριν την Διμερή Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και αυτό το ορόσημο είναι μόνο ένα μέρος από τις ε, ολαιόνα και στενότερες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Ε, επίσης, οι δηλώσεις αυτές αναφέρθηκαν στην ολοκλήρωση των, ε, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, μια συμφωνία που θα ολοκληρώσει τις ε, εμπορικές μας ε, σχέσεις. Η συμφωνία αυτή θα παρέχει μια πολύ ισχυρή βάση για την ε, περαιτέρω εξέλιξη της συνεργασίας μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, βιώσιμης ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και σε πολλούς άλλους τομείς. Η δήλωση αναφέρει ε, αναφέρθηκε επίσης ε, στην κοινή αντιμετώπιση κρίσεων και κοινά ψηφίσματα και τοποθετήσεις για ε, τις κρίσεις και δημιουργεί επίσης το πλαίσιο για τις διάφορες επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων που είναι κοινέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία. Αναφερθήκαμε επίσης στην ενίσχυση των θαλάσσιων επιχειρήσεων στο κέρας της Αφρικής και στον Ινδικό ωκεανό. Και η Αυστραλία θα εξετάσει τον ενδεχόμενο να στηρίξει και άλλες επιχειρήσεις ε, παρόμοιου τύπου. Επίσης, ε, στηρίζουμε τη δημιουργία ενός φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας που θα εμβαθύνει τις σχέσεις μας και τη διασύνδεση των ε, πολιτών μας. Η Αυστραλία τα τελευταία χρόνια σκοπεύει, προσπαθεί να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την περιοχή του Ειρηνικού αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνούμε τους ε, ε, ισχυρούς δεσμούς που έχουμε με την Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για διάφορα ζητήματα, για παράδειγμα γεωργικές ε, επιδοτήσεις, ε, τα τελευταία χρόνια οι διαφορές μας έχουν καλυφθεί από την ε, βαθύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας σε άλλους τομείς. Και αυτή η συνεργασία οφείλεται στο ότι μοιραζόμαστε κοινέ αξίες σε πάρα πολλούς ε, τομείς. Κάποια πρόσφατα παραδείγματα είναι ότι η Αυστραλία είναι ενωμένη με την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη στάση της ε, Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Και επίσης συμμεριζόμαστε ένα κοινό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια ζητήματα στην Ανατολική Ασία. Έχουμε τις ίδιες ε, προκλήσεις ε, σχετικά με την τρομοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ανταλλαγές ε, απόψεων και εμπειριών. Υπάρχει επίσης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλους τομείς που μπορεί να βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε όλο το ανεκμετάλλευτο δυναμικό στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας και ελπίζω σε μία ακόμα στενότερη συνεργασία έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε ε, ε, το στόχο αυτό συντομότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τέιλορ από την Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα και βλέπω φίλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αυστραλία. Είναι πολύ καλή η αφορμή να συζητήσουμε σήμερα την προτινόμενη εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία. Ο Υπουργός ο Αρμόδιος θα σταθεί στα θετικά και στα ωφέλη γενικότερα και για τις δύο πλευρές, αλλά θα ήθελα να σταθώ στα θέματα συνεργασίας από πλευράς μας και εταιρικότητας ε, όχι μόνο η συμφωνία αυτή θεωρεί ότι η περιοχή του Ειρηνικού, του Νότιου Ειρηνικού είναι μια κρίσιμη περιοχή για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η Νέα Ζηλανδία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο γι' αυτό. Εντυπωσιάζομαι γιατί βλέπω ότι η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια κοινή ανάγνωση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν και σε επίπεδο κλιματολογικών αλλαγών, και στα πλαίσια της αντιμετώπισης ε, κινδύνων ασφαλείας στην περιοχή του Ιράκ και της ε, ε, Συρίας και στην προσπάθεια επίτευξης μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού και για άλλα προβλήματα. Βλέπουμε ότι η δική μου χώρα προωθεί μια εμπορική συμφωνία πιο δίκαιη και πληρέστερη μάλλον με την Κίνα και με τις υπόλοιπες χώρες του ειρηνικού τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού. Σαν μέλος στην παρούσα φάση και του Συμβουλίου Ασφαλείας συμμεριζόμεθα τις απόψεις μας με τις υπόλοιπες χώρες και με τα μόνιμα μέλη ασφαλείας. Παρότι η ιστορία μας έχει φέρει σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο και θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε συμφωνίες που θα επηρεάσουν θετικά το μέλλον μας και την ανάπτυξή μας. Έχουμε πάρα πολλές συμφωνίες ήδη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες από άλλους και στον τομέα σαν παράδειγμα της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων. Μια νέα συμφωνία θα υπογραφεί το επόμενο έτος και θα έρθει και στο κοινοβούλιο σας ε, για επικύρωση. Έχει ολοκληρωθεί επίσης και η νέα συμφωνία της Τελωνιακής Ένωσης. Ε, συμφωνία για τις Τελωνιακές Συμφωνίες, συγγνώμη. Ε, η νέα εταιρική αυτή συμφωνία θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε πολύ στενές διμερός, διμερές, ε, θα έλεγα και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κι και ο Πρόεδρος Γιούνκερ ε, ε, αποφάσισα να προχωρήσουμε γρήγορα στην κατάληξη της διαδικασίας για την υπογραφή της νέας συμφωνίας. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε σαν Επιτροπή και σαν σύνολο Κοινοβούλιο όχι μόνο για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων αλλά για μια λύση ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές και μάλιστα να υπογραφεί και γρήγορα η συμφωνία. Ευχαριστώ και τους δύο πρέσβεις. Υπάρχει λοιπόν το πλαίσιο δεδομένο για την συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Μπορούμε να μπούμε σε βαθύτερο επίπεδο λεπτομέρειας. Θα ξεκινήσουμε με τη Νέα Ζηλανδία. 45 λεπτά για την Νέα Ζηλανδία. Θα συζητήσουμε μαζί τους λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εμπορική συμφωνία αλλά και τις ευκαιρίες. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες και μετά θα υπάρξει η δυνατότητα για κατάθεση ερωτήσεων προς τα μέλη. Πρώτον, χαίρομαι πράγματι που ο Υπουργός Εμπορίου της ε, Νέας Ζηλανδίας ε, είναι μαζί μας. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και για την αντιπροσωπεία της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας που βρίσκονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ήμουν βουλευτή στο παρελθόν και συνειδητοποιώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς πως έχουν τα πράγματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο προτού προχωρήσει διαπραγματεύσεις. Το όλο περιβάλλον των διαπραγματεύσεων έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα χρόνια. Και βλέπουμε πλέον ότι ε, η γενικότερη συνένεση σε ζητήματα εμπορίου έχει κάπως μετακινηθεί, έχει τροποποιηθεί και από ό,τι βλέπουμε είναι πλέον πολύ πιο σημαντικό για τους επαγγελματίες διαπραγματευτές να είναι σε επαφή με την πραγματικότητα σε κάθε χώρα, προκειμένου να κινείται προς σωστό χώρο και σωστή κατεύθυνση συζήτηση κάθε φορά. Εγώ για πρώτη φορά συμμετέχω σε συζήτηση στην Ευρώπη μετά τις αποτρόπες επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Γαλλία και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω στα γαλλικά. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπα στην ε, Comédie Française ε, στο Όκλαντ λίγη ώρα μετά τις τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις πρέπει να σας πω ότι εντελώς αυθόρμητα η γαλλική κοινότητα στο Όκλαντ δραστηριοποιήθηκε και αυτό που τους είπα είναι ότι μολονότι απέχουμε 15.000 ε, χιλιόμετρα από το Παρίσι, συμπονούμε απόλυτα τους πολίτες του Παρισιού και είπαμε ότι θα κάνουμε κάθε το δυνατό για να προασπίσουμε τον πολιτισμό μας. Πάση θυσία, πάση θυσία. Ήθελα απλώς να κάνω την παρέμβαση αυτή και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι πρέσβεις Χίγκη και Τέιλορ. Μιλάμε ουσιαστικά για κοινέ αξίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας. Είπαμε ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή κοινή ιστορία η οποία έχει αρχίσει να αποκρισταλώνεται όλο και περισσότερο μέσω του ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχουμε εφαρμόζονται μόνο σε έξι χώρες. Για όλες τις υπόλοιπες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντα μια προτιμησιακή διευθέτηση. Ενώ για τις έξι αυτές χώρες, Κίνα, Ταϊβάν, Ρωσία, Χονγκ Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ήταν χώρες οι οποίες δεν καλύπτονταν από συμφωνίες και αυτό φαινόταν κάπως περίεργο σε όλους εμάς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα των ε, βασικών αξιών που έθιξαν και οι δύο πρέσβεις. Θεωρώ και εγώ ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω της συμφωνίας αυτής να ευθυγραμμίσουμε περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές, εργασιακά δικαιώματα και πολλά άλλα ζητήματα που άπτονται του εμπορίου και των εργασιακών σχέσεων και από τις δύο πλευρές, Ευρωπαϊκή Ένωση και Νέα, Ζηλανδία. Πολύ σύντομα τώρα όσον αφορά το τομέα του εμπορίου. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το τομέα του εμπορίου καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματική μου ζωής και θυμάμαι μία μελέτη που έγινε το 2011 από 11, αν δεν κάνω λάθος, διεθνείς οργανισμούς με επικεφαλή στον ΩΣΑ όσον αφορά τη συνεργασία στα πλαίσια του ΠΟΕ, ILO και άλλων οργανισμών και ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν διάφορα αποδεικτικά στοιχεία από πολλές διαφορετικές εκατοντάδες μελέτες από τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν ε, ανοιχτές εμπορικές σχέσεις με πολλές άλλες χώρες όσον αφορά διάφορους τομείς. Το συμπέρασμα βασικά ήταν το ακόλουθο. Στις μελέτες εκείνες δεν υπήρχε καμία αρνητική επίπτωση από τις ε, ανοιχτές αυτές συμφωνίες εμπορίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις θετικές επιπτώσεις του εμπορίου, όχι να αναρωτόμαστε αν υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη διαπίστωση ότι οι ανοιχτέ ελεύθερες αγορές που συνεργάζονται επιφέρουν και θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τη Νέα Ζηλανδία, ε, είμαστε η 52η μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε περίπου 150 οικονομίες που είναι μικρότερες από, τη δική, από την δική μας. Επομένως, μπορούμε και εμείς ως μικρή αλλά ενδιαφέρουσα για την Ευρώπη αγορά να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο. Ένα στατιστικό δεδομένο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεδομένης της έμφαση της Νέα Ζηλανδία στο γεωργικό τομέα. Τα τελευταία πέντε χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πηγαίνουν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας και βλέπουμε ο μέσος όρος ανάπτυξης του κλάδου αυτού, των εξαγωγών μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Νέα Ζηλανδία, είναι 20% σε τήσια βάση. μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Νέα Ζηλανδία και αυτό πρόκειται να αυξηθεί. Ξέρετε ότι στον γύρο της Ουρουάης είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για τις σχέσεις που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα τότε ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπήρχαν κάποιες ρήτρε τις οποίες θεωρούσαμε ιδιαίτερα ευαίσθητε και έπρεπε πάση θυσία να τηρήσουμε, αλλά βλέπουμε πλέον ότι όσον αφορά συγκεκριμένου τομεί όπω τα γαλακτοκομικά προϊόντα, βλέπουμε ότι οι ε, εξαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία προς το εξωτερικό έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά γαλακτοκομικά πλέον προϊόντα τα οποία εξάγουμε με πολύ πιο έντονους ρυθμούς από τη Νέα Ζηλανδία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί η Κίνα και οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν αλλάξει εντελώς το περιβάλλον, το τοπίο όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξάγουν πολλά γεωργικά προϊόντα, όπω ξέρετε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλέ πλέον επιχειρήσει τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίε επενδύουν στον γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύσει σε γαλακτοκομικέ επιχειρήσει εδώ πέρα στην Ευρώπη και βλέπουμε πλέον ότι ε, οι επενδύσεις όλο και διαφοροποιούνται. Επομένως έχουμε επενδύσεις και σε άλλους τομείς θα μπορούσα να αφαιρθώ σε κάποιους ε, στρατηγικούς τώρα προσανατολισμούς όσον αφορά τον ρόλο που έχουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πολύ θετικά εν ώψη της Συνόδου του Ναϊρόμπι. Βλέπουμε ότι ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών η Νέα Ζηλανδία έχει προσπαθήσει να συμβάλλει σε αυτές τις συμφωνίες. Είναι όσον αφορά το TPP για παράδειγμα ένας από τους θεματοφύλακες στη Νέα Ζηλανδία. Ξέρετε ότι καταφέραμε να συνάψουμε πρόσφατα αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέση των χωρών του Ειρηνικού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις αρχικές μου παρατηρήσεις, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Έχει οριμάσει πλέον η διαδικασία, είναι σίγουρα πολύπλοκη, δεδομένου ότι συμμετέχουν 28 κράτη-μέλη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε τελικά να έχουμε μία συμφωνία του 21ου αιώνα πλέον που θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών και στις δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ο δεύτερο εμπειρογνώμονα για την Νέα είναι ο κύριος Μακιγιάμα και έχετε αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητέ κύριε Υπουργή. Με μεγάλη μου χαρά παίρνω τώρα το λόγο μετά από τους εκλεκτούς ε, καλεσμένους πρέσβεις. και μετά μάλιστα από την ε, υπογραφή της συμφωνίας TPP που έγινε τον ε, περασμένο μήνα. Είναι προφανές ότι η TTP είναι, θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην οποία δεν θα συμμετέχει η Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο, ε, μεγαλύτερη συμφωνία τέτοιου είδους μετά από τον γύρο της Ουρουγουάης και τα αποτελέσματα αυτής της, συμφωνίας θα γίνουν αισθητά. Και στις ε, χώρες ε, TPP υπάρχουν μόνο δύο οι οποίες ε, δεν συμμετέχουν. Δεν έχουμε άλλο, άλλη επιλογή από το να συμμετέχουμε όλοι στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να διαπραγματευτούμε αυτές τις δύο συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Βέβαια, το ενδιαφέρον για την πρόσβαση στην αγορά και της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας είναι κάτι πολύ ελκυστικό. Μιλάμε για ένα τυφλό σημείο που ανέρχεται στο 1,5-3 εκατομμύριο αμερικανικά δολάρια. Η Αυστραλία είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, όμως και τα και η Νέα Ζηλανδία έχει μεγαλύτερο ε, ΑΕΠ από εκείνο του Περού και του Βιετνάμ με, με τις ε, οποίες χώρες κοντεύουμε να συνάψουμε τις ε, συμφωνίες που γνωρίζετε. Όσον αφορά την κατανάλωση, είναι μια οικονομία η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη της Μαλαισίας, της Χιλής και της Σιγκαπούρης. Δηλαδή, ε, το δυναμικό της ε, αγοράς, ιδιαίτερα των εξαγωγών μιας οικονομίας όπως της Νέας Ζηλανδίας, είναι πολύ μεγαλύτερο από Τη οικονομίες των χωρών που ανέφερα. Γι' αυτό είναι προ το συμφέρον όλων να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Εάν δηλαδή μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με την Σιγκαπούρη, τότε με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε ήδη να έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσει με τη Νέα Ζηλανδία. Και συνεχίζοντα από αυτό να πω ότι ακούσαμε ήδη για το ε, πόσες υπάρχουν, ε, πόσο μεγάλο είναι το επίπεδο συνοχή και πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτά μιλώντας για την ε, τίτη. Και προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την ε, συμφωνία TTIP, είχαμε μόνο δύο συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης σε ισχύ. Με τις υγείες σας για τις ε, τηλεπικοινωνίε και τον εξοπλισμό και για τα σκάφη πολυτελεία. Είχαμε καλύψει όλους τους, τομείς, ε, τους μεταποιητικούς τομείς και ε, το SPS. Είναι μία άνευ προηγουμένου φιλόδοξη προσπάθεια και πολλές φορές αναφερόμαστε ανεπίσημα σε αυτή ως μία συμφωνία ιστορική. Φυσικά, τα πρότυπα ασφάλειας των ετροφίμων στη Νέα Ζηλανδία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ακούσαμε επίσης ε, τα σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους και να σας πω πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό και για τις εξαγωγές στην Ευρώπη και μάλιστα στα πλαίσια του πολιτικού κλίματος και της αυξανόμενης ευαισθησίας των Ευρωπαίων πολιτών προς την προστασία των ε, δεδομένων. Δεν θέλουμε να ε, θέσουμε σε κίνδυνο την ακαιρεότητα και την ελευθερία μας και αυτό είναι ένα τομέας στον οποίο μπορούμε να ε, δράσουμε και να συζητήσουμε το θέμα των ροών δεδομένων. Επίσης, ε, το θέμα της αγιοργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, όπως πολύ σωστά ε, αναφέρεται, είναι εξαγωγή γεωργικών προϊόντων. Και είναι μεγάλη ε, εξαγωγή. Και όλες οι χώρες, με εξαίρεση την Σιγκαπούρη, αν δεν κάνω λάθος, εξάγουν γεωργικά προϊόντα. Το ύψο των εξαγωγών αυτή τη στιγμή της Νέας Ζηλανδία ανέχεται στα 60 δισεκατομμύρια, στα 26 της Αυστραλίας στα 30 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 67 δισεκατομμύρια. Το μερίδιό μας είναι μικρό σχετικά, όμως καθόλου ομεληταίο. Ε, δεν θα αναφερθώ στον γεωργικό τομέα της Αυστραλίας, αυτό θα το ε, αναπτύξουν περισσότερο οι άλλοι καλεσμένοι. Όμως ε, για την Νέα Φιλανδία να σας πω ότι τα προϊόντα που εξάγουν είναι ε, ως ε, επιτοπλίστων χωρίς δασμούς. Μιλάω για κτηνοτροφία, για ζώα, για πρόβατα, για βούτυρο, βοδινό κρέας και τα προϊόντα ε, τα οποία ακόμα έχουν δασμούς ε, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ε, με τα προϊόντα του βόρειου ημισφαιρίου. Μιλάμε για προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται σε άλλες εποχές του χρόνου. Και οι εξαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία μας επιτρέπουν να έχουμε στη διάθεσή μας όλο τον χρόνο ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Ε, τώρα, εξάγουμε επίσης ε, κρασί, όμως και εδώ υπάρχει μεγάλη ε, επικάλυψη. Η Νέα Ζηλανδία εξάγει κρασί και εξάγει κρασί της ποιότητας Sauvignon Blanc, να σας πω. Τώρα δεν θα αναφερθώ στον γαλακτοκομικό τομέα θα αρκεστώ στο να πω πως ε, είμαστε πάρα πολύ ε, ανταγωνιστικοί. Όμως η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης ανταγωνιστική. Ε, βέβαια, μην ξεχνάμε και το θέμα της απόστασης. Η απόσταση είναι απαγορευτική για να εξάγει η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα μάλλον προς την Ευρώπη. Χρειάζονται 32-33 μέρες για να φτάσει ένα πλοίο από την Αυστραλία στην Ευρώπη. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιος ε, κίνδυνος. Τώρα, από τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει, έχουμε εντοπίσει κάποιες ευαισθησίες που πιστεύω πως οδηγούν σε φόβους που δεν είναι βάσιμοι. Είμαστε οικονομίες διαφορετικού μεγέθους. Και υπάρχουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες στον γεωργικό τομέα και σε κάποιους ε, άλλους τομείς, ε, όπως για παράδειγμα την, ε, τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να δημιουργήσουμε τη νέα ε, γενιά ε, μιας συμφωνίας η οποία θα φροντίζει τόσο το συμφέρον της ε, Ευρώπης όσο το συμφέρον των χωρών μας. Και πιστεύω πως είναι το κατά, η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αρχίσουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια τέτοια συμφωνία. Σίγουρα καμία διαπραγμάτευση δεν είναι ανώδυνη, όμως για να είμαι ειλικρινής, εάν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Νέα Ζηλανδία, νομίζω πως δεν θα καταφέρουμε να ε, διαπραγματευτούμε με καμία άλλη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος εμπειρογνώμων είναι ο κύριος Πέσονεν, Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠΑ. και ειδικό σε θέματα γεωργίας. Και μια που η γεωργία είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα, θα σας δώσω αμέσω στο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Με χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Θα σας δώσω κάποιες από τις σκέψεις τις οποίες κάνει η κοινότητα η αγροτική στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων των οικονομικών με ε, τους συναδέλφους από τους αντίποδες. Εμείς βλέπουμε ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη απασχολούνται άμεσα στην ε, γεωργική δραστηριότητα μαζί με άλλους βέβαια έμεσα φτάνουμε τα 40 περίπου εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ο μεγαλύτερος αν θέλετε εργοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρωσική κρίση άλλαξε την κατάστασή μας με δραματικό τρόπο. Έπρεπε να επιλέξουμε διαφορετικές λύσεις σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Ξεκίνησαν πρωτοβουλίες για διαφορετικές αναλλακτικές εμπορικές πρακτικές για να καλύψουμε τις ανάγκες και αυτό είναι που μας απασχολεί στην παρούσα φάση. Είδαμε ότι το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής υπήρξε μια αύξηση 6,7% των γεωργικών προϊόντων, της παραγωγής και των συναλλαγών αλλά ε, με χαμηλές τιμές αγοράς των προϊόντων και ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετώπισαν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς όπως το, βόλιο, το χείριο συγγνώμη, κρέας και ε, η γαλακτο, γαλακτοκομία. Ε, με τη Νέα Ζηλανδία συνδεόμεθα σε τομείς πολύ στενά όπως η γαλακτοκομία έχουμε πολλούς κοινούς παρανομαστές θα έλεγα στα πλαίσια της του εμπορίου γεωργικών προϊόντων με την χώρα αυτή, καζεΐνη, αποκορυφωμένα γάλατα και γενικά υπάρχει συνεργασία και σε, ε, στις υπόλοιπες περιοχές του Ειρηνικού και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εγώ συνάντησα εδώ στις Βρυξέλλες ε, κάποιους εμπειρογνώμονες ε, μαζί με τους δύο συμπροέδρους της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ και το εμπόριο είναι ε, ένας δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Είναι αμφίδρομη η σχέση την οποία θα πρέπει να έχουμε και να παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους. Η Νέα Ζηλανδία είναι ένας πολύ καλός σύντροφος και σύμμαχος. Έχουμε καλές επαφές με τους συναδέλφους μας, συναντώμεθα με τους εκπροσώπους της Γεωργίας από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία Έχουμε τακτικές επαφές σε τομείς όπως την παραγωγή προβίου κρέατος και το χείριο επίσης. Υπάρχουν αρκετές διαφορές, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, η απόσταση ανάμεσα σε εμά και στη Νέα Ζηλανδία, αυτό υπόθηκε και από τους προηγούμενους βέβαια ομιλητές. Όμως, ε, όπως είπε και ο κύριος Κρόζερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους αριθμούς μου στέλνει προϊόντα που ξεπερνούν σε ετήσια βάση τα 750 εκατομμύρια και εισάγουμε ε, περίπου 2 δις προϊόντα γεωργικής, γεωργικά αξίας άνω των 2 δις. Υπάρχει δηλαδή μια ανισορροπία. Θα ήθελα να πω επίσης και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το TTP Υπάρχουν δύο πλευρές ε, που απασχολούν τη γεωργική βιομηχανία και τις συνεστερητικές οργανώσεις. Εμείς έχουμε μια ευνοϊκή γενικά θέση σε ορισμένες αγορές όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και έχουμε μια καλή πρόσβαση, έχουν οι Νεοζηλανδοί μια καλύτερη από εμά πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές εις βάρος των ευρωπαϊκών. Ανησυχούμε λοιπόν για τα μειονεκτήματα τα οποία δημιουργούνται για τους παραγωγούς μας σε χώρες όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά από τη συμφωνία, μετά τη θέση σε ισχύ τη συμφωνία TPP. Να υπογραμμίσω επίσης ότι μιας και ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος και το μέγεθος της οικονομίας γενικότερα είναι σημαντικός. Έχουμε διαφορές. Υπάρχουν τομείς όπως η αλλακτοκομία ε, και τα οποροκυπευτικά που κυριαρχούν την οικονομία και κυριαρχούν στο εμπόριο ανάμεσα στην Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία. Ενώ στη δική μας περίπτωση στην ενιαία αγορά ο ρόλος των συγκεκριμένων αγορών αυτών είναι πολύ χαμηλότερος. Εκτιμούμε πάντως την διαθεσιμότητα των εμπορικών μας εταίρων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το πρόβιο κρέας, αλλά υπάρχουν ανοιχτά θέματα και όταν μιλάμε για προϊόντα με προστιθέμενη αξία, αυτά θα επηρεάσουν νομίζω στο μέλλον τη ζωή των γεωργών και κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους αυτούς τομείς, δηλαδή γαλακτοκομία και παραγωγή βοήου και πρόβειου κρέατος. Λοιπόν, θα ήθελα στις διαπραγματεύσεις να υπάρξουν κάποιες ε, σημαντικές προόδοι, ιδιαίτερα σε σχέση με την εποχικότητα και άλλα θέματα. Τώρα για τα μη δασμολογικά. Η Νέα Ζηλανδία θεωρείται ότι έχει υψηλού επίπεδο προστασία της αγοράς της απέναντι στις ε, εισαγωγές δόθηκαν κάποια παραδείγματα σύμφωνα με τις δικές μας στατιστικές το ποσοστό της αγοράς ε, στα μήλα σαν παράδειγμα είναι ε, ασήμαντο παρά το ότι εισάγουμε πολλά μήλα από τη Νέα Ζηλανδία όταν μιλάμε δηλαδή για την εποχικότητα ε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είναι αμφίδρομη η σχέση και δεν είναι τώρα σε σχέση με τον κτηνιατρικό και, φυτο, και τον έλεγχο των, της φυτικής παραγωγής εμείς θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωριστεί σαν μια ενιαία οντότητα ε, δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα από πλευρά των Νεοζηλανδών και βέβαια δεν είναι ο χειρότερος σε εισαγωγικά πελάτης η Νέα Ζηλανδία. Έχουμε ε, κάποια θέματα πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια των οποροκυπευτικών. Τα ακτινίδια σαν παράδειγμα θα θέλανε και τα δικά μας προϊόντα να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην νεοζηλανδική αγορά. Ε, τώρα για τα προϊόντα γεωγραφικής ελεγχόμενης προέλευσης. Νομίζω ότι για μας, για αυτά τα προϊόντα, τα λεγόμενα GI, η γεωγραφική ένδειξη έχει κάτι το πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Με αποτελεσματικά οικονομικό τρόπο μας επιτρέπει να οργανώσουμε την παραγωγή προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη. Θα θέλαμε η Νέα Ζηλανδία να αναγνωρίσει αυτή την αρχή όπως το κάνει και ο Καναδάς. και αυτό θα οδηγήσει στην παραγωγή και την προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με τη Νέα Ζηλανδία αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το να φέρουμε σε επαφή τους αντίστοιχους τομείς στη Νέα Ζηλανδία με τον πολυτομεακό τρόπο ε, που αντιμετωπίζονται τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχουν οι ευρωβουλευτέ. Δύο έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο. κύριο Φέλνερ, Κέλλη και Χάιντσον. Λοιπόν, καταγράφουμε τα όνοματά σα. Φέλνερ πρώτος. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Καταρχάς, σα ευχαριστώ για τις εξαιρετικέ αυτές παρουσιάσεις. Είναι πολύ θετικό να ξεκινάμε με τόσο επικοδομητική ατμόσφαιρα τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ εύκολα όταν ακούμε τους εμπειρογνώμονε ε, σε σχέση με άλλες διαπραγματεύσει που χρειάστηκε να διεξάγουμε. Ένα σημείο που μας είχε απασχολήσει και με τον κύριο Ντιμαρτή και ο Ντέβιτ Μάρτιν επίσης το είχε δει ε, αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλές ε, υποδιαπραγμάτευσεις συμφωνίες και προσθέτουμε και άλλες συνεχώς. Το σημαντικό είναι να μην ξεκινάμε μόνο, αλλά και να ολοκληρώνουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ. Μία ερώτηση απίθανη λοιπόν. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τις δύο αυτές συμφωνίε. Σε ένα χρόνο, σε πόσο καιρό θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις συμφωνίες. Και όταν έθεσα το ερώτημα αυτό στο παρελθόν, τελικά διαψεύστηκα. Πιστεύετε ότι έχουμε ένα φιλόδοξο και παράλληλα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τις δύο αυτές συμφωνίες. Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρουσιάσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε στο TPP και είπατε ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τη Νέα Ζηλανδία, ιδίως όσον αφορά τις εξαγωγές στις προς Πολιτείες. Αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το TTIP, δεν πιστεύετε ότι αυτό θα αντισταθμίσει και ενδεχομένω να επηρεάσει την εφαρμογή της TPP. Μήπως θα έπρεπε και για αυτόν το λόγο να επιταχύνουμε την σύναψη της TTIP με τις ΗΠΑ. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η μέση τάξη διωγγώνεται όλο και περισσότερο στο Βιετνάμ, την Ινδονησία, γενικότερα στην Ασία, η μεσαία τάξη. Δεν θα έπρεπε να κληθεί η Νέα Ζηλανδία να καλύψει αυτή τη νέα αναδυόμενη αγορά. Γιατί θέτουν αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή αγορά ως προτεραιότητά τους, αλλά λάβουμε υπόψη την τεράστια απόσταση που διαχωρίζει την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία από την Ευρώπη, θα ήταν πιο ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ασιατική μεσαία τάξη. Και τρίτον, η Ιρλανδία ξέρετε ότι είναι και αυτή γεωργική χώρα, εξαρτάται πάρα πολύ από τις εξαγωγές, 80% του ΕΠ μας προέρχεται από τις εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διαπραγματεύσεις στις οποίες θα πρέπει να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις όσον αφορά το γεωργικό τομέα και τον κτηνοτροφικό τομέα. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας, Κάσπαρη. Πολύ συχνά οι Ευρωπαίοι πολίτες μας λένε ότι έχουμε πολλά αμυντικά συμφέροντα, το ίδιο και οι εταίροι μας. Και εγώ τους εξηγώ ότι όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αμυντικά συμφέροντα έχει και άλλη πλευρά, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως μπορούμε να βρούμε λύσεις. Τα δικά σας τα αμυντικά συμφέροντα ποια είναι. Ποιους κλάδους θέλετε να προστατεύσετε προς τον κύριο Πέσονεν. Είπατε ότι υπάρχει μία ανισορροπία όσον αφορά τα εποχικά αυτά προϊόντα, τα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται από μία κάποια εποχικότητα. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Εγώ πίστευα ότι θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Έχουμε τα ίδια προϊόντα και διαφορετικές εποχές, άρα θα ήταν εύκολο να εξάγουμε ή να εισάγουμε τα προϊόντα αυτά. Θα υπήρχε μια συμπληρωματικότητα. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν πού έγκυται το πρόβλημα. Ναι, έχουμε διαφορετικά πρότυπα, διαφορετικέ προδιαγραφέ, αλλά για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η εποχικότητα των προϊόντων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Ευχαριστούμε, ο Ντέιβιντ. Σα ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που βλέπω εδώ και τον Υπουργό και του υπόλοιπους καλεσμένους. Ξέρω ότι σημειώνεται πρόοδος ε, για τις δύο αυτές συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες αυτές το συντομότερο δυνατό. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αντίθετη από αυτή που έκανε ο Ντάνιελ. Σε ποια σημεία η Νέα Ζηλανδία έχει επιθετική στάση. Καταλαβαίνω ότι ο γεωργικός τομέας θα είναι ενδεχομένως ένας από τους τομείς όπου η Νέα Ζηλανδία θα έχει μια πιο επιθετική στάση. Τι έχει να κερδίσει ουσιαστικά η Νέα Ζηλανδία από την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική της Νέας Ζηλανδίας και απευθύνομαι κυρίως στον Υπουργό Επορίου. Ξέρετε ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τα γενικότερα μέσα τα οποία είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες, όπως για παράδειγμα το ISDS ή κάποια άλλα στοιχεία, νομίζω ότι αντίστοιχα θέματα πρέπει να υπάρχουν και στη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή θέματα επί των οποίων ενδεχομένω να, να σταματήσει όλη η διαπραγματευτική διαδικασία. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα καθόδη ζητήματα για σας. Ευχαριστούμε. I'm also pleased. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ πέρα τους καλεσμένους μας, καθώς επίσης και τον Υπουργό Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας. Πολύ θετικέ, πολύ καλές ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Να πω και εγώ με τη σειρά μου κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει για τη σύναψη μια εμπορική συμφωνία. Έχουμε κοινέ αξίε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και στον τομέα του εμπορίου να αντικατοπτρίζονται οι αξίες αυτές όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θέλω όμως να ξέρω πιο συγκεκριμένα τι έχει να κερδίσει η Νέα Ζηλανδία από τις διαπραγματεύσεις αυτές, ποια είναι η ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τη Νέα Ζηλανδία. Και ξέρω ότι ενδεχομένως στο στάδιο αυτών των διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως να έχετε κάποιους κρυμμένους άσους. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω η δική σας η επιθετική πολιτική ποια θα είναι στα πλαίσια πραγματεύσεων. Ποιους τομείς θέλετε να προασπίσετε. Κύριε Κράσφαντερ Χάινς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για αυτήν την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε. Έχω μια ερώτηση με τον κύριο Χιμαγιάμα. Έχουμε διάφορες εμπορικές συμφωνίες και όντως είμαστε σε στάδιο διαπραγματεύσεων για ε, πολλές από αυτές. Μια ερώτηση λοιπόν προς ε, την Κομισιόν. Υπάρχουν ε, οι διαθέσιμοι πόροι για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Και μιλώ για τους διαθέσιμους πόρους όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις αλλά και για την εφαρμογή των συμφωνιών. Και όπως είπε και ο κύριος Κασπάρη, για τον κύριο Πεσόνεν, η πρόσβαση στην αγορά είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ε, δεν υπάρχει μήπως κίνδυνος να ε, η αγορά από διάφορα προϊόντα από αυτές τις χώρες ή για παράδειγμα από ακτινίδια. Ε, δεν πρέπει να προσέξουμε και αυτό στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνουν στο τέλος και των δύο ε, συζητήσεων με τα δύο πάνελ δεν έχει κάποια σχέση αυτή με τους επιδεγνωμόνες. Ο κύριος Περέιρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους ε, προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτα στον Υπουργό Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας ε, για την TPP, τη συμφωνία TPP. Η χώρα σας φυσικά είχε πολύ έντονες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από ε, τις διαπραγματεύσεις. Διδάγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ε, στις δικές μας διαπραγματεύσεις. Ποια είναι η δική σας οπτική γωνία για την ε, συμφωνία ανάμεσα στην Νέα Ζηλανδία και τους εταίρους της συμφωνίας TPP και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και μια άλλη ερώτηση που έκανε ήδη ο David Μάρτιν σε σχέση με τους επενδυτές, την προστασία των επενδύσεων. Όπως ξέρετε στην Ευρώπη συζητούμε έντονα αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια πρόταση για ένα επενδυτικό δικαστήριο. Το... Έχουμε επίσης και το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτου, το ISTS. Θα ήθελα να μάθω για την δική σας οπτική γωνία. Μήπως ε, έχετε κάποια εναλλακτική την οποία ε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε ή θεωρείτε πως ε, η συνηθισμένη επίλυση διαφορών είναι η καλύτερη επιλογή. Κύριος Ντάρτμαουθ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω καταρχάς ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μια συμφωνία ελεύθερου με τη Νέα Ζηλανδία και της γυρίσαμε την πλάτη το 1973 έως το 1975 και 40 χρόνια αργότερα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά μια τέτοια συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. Και φυσικά άλλο να το συζητάμε και άλλο να το δούμε να εφαρμόζεται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και σας παρακαλώ ε, να μην θεωρήσετε πως είμαι επιθετικός απέναντί σας. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Η τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή ε, ξοδεύουμε τον περισσότερο χρόνο που έχουμε συζητώντας αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό δηλαδή που θέλω να ρωτήσω είναι, δεδομένων αυτών, τι περιμένετε εσείς να αλλάξει με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεδομένου ότι υπάρχει μια συμφωνία τέτοια ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και την Κίνα, ποια είναι η διαφορά που έκανε αυτή η συμφωνία στο εμπόριό σας με την χώρα αυτή και τι αναμένετε ποσοτικά. Τι θεωρείτε εσείς πως θα καταστήσει μια ικανοποιητική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ. Καταρχά να ζητήσω συγγνώμη που έλειπα στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, αλλά να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι συζητάμε εδώ την συμφωνία αυτή με την Αυστραλία και τη Νέα Συλλανδία που όπως ε, ακούστηκε ήδη είναι χώρες που συμμερίζονται κοινέ αξίες με εμάς. Οι δικές μου ερωτήσεις είναι για τους ε, υπουργούς. Ποιοι είναι οι κοινοί μας στόχοι, τι μπορούμε να επιτύχουμε, ποιες ε, είναι οι δυνάμεις που μπορούμε να ενώσουμε και πώς μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο ταχύτερα για τις διαπραγματεύσεις. Και κάτι άλλο που με απασχολεί αρκετά. Ε, μιλούμε για το εμπόριο για όλους και το πώς ερμηνεύει ο καθένας μας αυτήν την φράση. Ε, τι σημαίνουν οι εμπορικές συμφωνίες για τους απλούς πολίτες, ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχουν στις καθημερινές τους ζωές. Βλέπω πως ε, δυσκολεύεστε να αναφερθείτε στα ωφέλη της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου εμπορίου και ίσως θα μπορούσατε να μας ε, πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Έχετε τέσσερα λεπτά ο καθένας για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά για όλες αυτές τις ερωτήσεις θα απογοητεύσω κάποιους από εσά, πολλούς από εσά, δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσω με επάρκεια. Να αναφερθώ σε αυτά τα οποία θέσατε γενικότερα σαν θέματα για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και την ταχύτητα. Κοιτάξτε, το ταχύτερο δυνατόν. Εμείς μπορούμε να, να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε με την ταχύτητα και την οποία εσείς μπορείτε να έχετε από πλευρά σας είναι μια διαδικασία περίπλοκη γιατί πρόκειται για 28 μέλη. Εμείς μπορούμε να πάμε γρήγορα. Τώρα για την καταλληλότητα ε, των πόρων της, ε, των διαπραγματευτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έχουμε συζητήσει αναλυτικά με εκπροσώπους υψηλού επίπεδου που γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν βλέπω να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αλλά αυτό είναι κάτι που άπτεται της αποτελεσματικότητας της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Θα μπορούσαμε να τα διαπραγματευτούμε αυτά με εξαιρετική ταχύτητα. Κάποια άλλα θέματα στα σχόλια σας, γιατί η Νέα Ζηλανδία θέλει να το κάνει ε, και γιατί θεωρεί ότι έχει συμφέρον να το κάνει με την Ευρώπη. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Για μας είσαστε μια πάρα πολύ σημαντική αγορά. Ε, πολύ λιγότερο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν. Η Νέα Ζηλανδία στην ουσία ήταν, είχε δημιουργηθεί σαν ένα αγρόκτημα offshore του Ηνωμένου Βασιλείου και το 60% των εξαγωγών μας μέχρι πριν λίγο καιρό πήγαιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε όταν θέτετε αυτήν την πολύ λογική ερώτηση γιατί ενδιαφέρεστε για την Ευρώπη και δεν θα ήταν καλύτερα για σας να στραφείτε στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η απάντησή μας είναι σαφής. Η διαφοροποίησή μας σε σχέση με τις αγορές ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική. Οι εμπορικές μας συμφωνίες έχουν πάει πάρα πολύ καλά και οι συμφωνίες που ήμουν, μάλιστα ήμουν εγώ εκπρόσωπος της Νέας Ζηλανδίας στην Ουρουάη, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε εκπληρώσει τις ποσοστώσεις που είχαμε για το πρόβιο κρέας 222.000 ε, τόνους σε κάποια φάση για χώρες όπως η Κίνα. Λοιπόν, ε, στο, στο πρόβιο κρέας δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Για το βούτυρο στα γαλακτοκομικά ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα και έτσι και αλλιώς ε, η ευρωπαϊκή αγορά τυρού φτάνει τα 4 εκατομμύρια τόνους. Οπότε εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική εξαγωγική δυναμική. Και δεν θέλουμε να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ε, στα πλαίσια από τις συμφωνίες στις προτιμησιακές τις οποίες έχει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με φίλους και ανταγωνιστές. Θέλουμε απλά να υπάρχει ισοτιμία σε σχέση με κάποια από τα υπόλοιπα θέματα. Το ISDS είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Στην ουσία είναι η βασική πολιτική ανησυχία στη χώρα μου και κατανοώ και το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά του, του αν θέλετε του λάκου σε εισαγωγικά που μας χωρίζει και όταν αναφέρομαι σε λάκο αναφέρομαι στη θάλασσα που μας χωρίζει από την Αυστραλία 1200 μίλια απόσταση. Ε, και υπάρχουν λοιπόν κάπως, ε, κάποιες ανησυχίες, προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τις αγορές λέγοντας ότι εμείς σε σχέση με το ISDS δεν έχουμε μια δεδομένη άποψη. Εμείς βλέπουμε το τι κατετίθεται σαν πρόταση, υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες και αν είναι επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουμε για κάποια νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή, γιατί όχι, σχετικά με τα GI, τη γεωγραφική προέλευση, ένδειξη. Ε, πρέπει να νομίζω και αυτά τα οποία από εκπρόσωπος της ΚΟΠΑΚΟΖΕΚΑ τα κατανοούμε πλήρως και μπορούμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε έτσι ώστε να μην διαταράξουμε ε, την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ μακριά από πουδήποτε, είμαστε η πιο απομονωμένη χώρα στον κόσμο, δεν έχουμε ασθένειες ενδυμικές σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το SPS ε, και τον υγειονομικό έλεγχο με βάση επιστημονικές μελέτες. Έχουμε ένα ειδικό ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα προστασίας και είμαστε διατεθειμένοι να το επανεξετάσουμε. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις, επαναλαμβάνω, μετακινούμεθα. Εμείς είχαμε πάρα πολλές αρνητικές στάσεις γύρω από αυτό. Εγώ προσωπικά δεν ήμουνα υπέρ αυτών των αντιστάσεων γιατί νομίζω ότι τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα τερουάρ όπως λέγονται ε, ε, μπορεί κανείς να δείξει κατανόηση, δεν πρέπει να είναι απόλυτος. Άλλωστε ξεκινήσαμε και εμείς με κάποιους νέους κανονισμούς ε, για ένα κατάλογο, ένα μητρό γεωγραφικών ενδείξεων και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αλλά δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτό. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω επαρκώς όλες τις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι το εξής. Δεν είναι τόσο δύσκολη η ιστορία. Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο να το κλείσουμε το θέμα και θα το κάνουμε με αποτελεσματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λί Μακιγιάμα. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε και όλα αυτά τα οποία είπατε σε μια συνέντευξη του 2014. Δεν ξέρω σε τι να φέρεστε ακριβώς κύριε Πρόεδρε, πάντως ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εγώ είμαι φύση απεσιόδοξος και πολύ συχνά έχω δίκιο τελικά όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά όμως τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, όσον αφορά τη δυνατότητα επίτευξη συμφωνίας, ναι, αυτή είναι πολύ υψηλή. Όσον αφορά όμως το χρονοδιάγραμμα, εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, ιδίως όσον αφορά τη Νέα Ζηλανδία, διότι Πρώτον, το ζήτημα που τίθεται δεν είναι να προχωρήσουμε αναγκαστικά γρήγορα ως διαπραγματευτές, αλλά κυρίως να δούμε πώς θα αναλώσουμε τον χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Από όσο καταλαβαίνω, η Νέα Ζηλανδία δεν διαπραγματεύεται βάση συγκεκριμένου πίνακα. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε έναν πόλεμο χαρακτή σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε εντελώς διαφορετικές συζητήσεις. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε όχι πόσο χρόνο θα χρειαστεί να διαπραγματευόμαστε, αλλά πώς θα διαπραγματευόμαστε. Τώρα, αν αξίζει να ταπανίσουμε όλο αυτό το χρόνο και όλου αυτού του σπόρου, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων, πιστεύω. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές, ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες εξαρτώνται από τις εξαγωγές. Ακόμα και η Γαλλία αυτή τη στιγμή εξαρτάται περισσότερο από τις εξαγωγές από ότι η Κίνα. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπορική εξάρτηση παγκοσμίω, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών είναι να δημιουργήσουμε συμφωνίες που καλύπτουν όλο αυτό το πολυμερές πολύπλοκο περιβάλλον και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να διασώσουμε, θέλετε, το δικό μας μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε οικονομίες εξαγωγών όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Ας περάσουμε τώρα στο TTIP. Το 2008 όταν έγινε η πρώτη αυτή πρόταση για, την, για το TTIP, πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι εντελώ τρελό να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Πολλοί εξακολουθούν και το πιστεύουν. Παρ' όλα αυτά, η TTIP δεν αποτελεί πανάκια, δεν πρόκειται να λύσει όλα μα τα προβλήματα. Ιδίω για κάτι που ισχύει εδώ και 10 χρόνια. Ότι το κέντρο πλέον του οικονομικού κόσμου έχει μετακινηθεί προ την Ασία και τον Ειρηνικό. Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε συνειδητοποιούν πλέον ότι το μέλλον του δεν διαμορφώνεται τόσο πολύ στα πλαίσια τη ε, TTIP. Έχουν τεθεί κάποιες βασικές πολιτικές προτεραιότητες, αλλά δυστυχώς σταματήσαμε εκεί στα πλαίσια του TTIP. Πολλές φορές βλέπουμε ότι όσον αφορά την ε, παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, αν δεν έχουμε το TTIP, δεν θα έχουμε και καμία ισχύ τελικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν παράλληλα και το TPP, δεν βασίζονται μόνο στο TTIP. Επίσης, μέσω του TTIP θα κερδίσουμε μεγάλα ποσοστά όσον αφορά το ΑΕΠ μας. Αν επικυρωθεί λοιπόν η TTIP, θα καταφέρουμε να επανέλθουμε σε μία κατάσταση η οποία θα είναι αποδεκτή, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να σημειώσουμε πρόοδο και να μετράμε περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, θα χρειαζόμαστε και άλλε συμφωνίε, όπω αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Ακούσαμε ότι εξάγουν πάρα πολλά προϊόντα προς την Ασία και τον Ειρηνικό, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Βέβαια δεν τις κατακρίνουν για κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί πέρα μπορούν τελικά να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη ενδεχομένως να πρέπει να θέσουμε την ευρωπαϊκή αυτή συμφωνία που θέλουμε να συνάψουμε τις δύο αυτές χώρες σε έναν άλλο περιβάλλον. Ενδεχομένως να μην θέλουν να εξάγουν ακόμα περισσότερα προϊόντα σε εμά, αν δούμε για παράδειγμα την περίπτωση τη Νέα Ζηλανδία. Έχουν ε, καλύτερο καιρό από πολλές χώρες, από την Εστονία για παράδειγμα, αλλά οι αρωτρέ εκτάσει που παραμένουν ακόμα για τη χώρα αυτή ουσιαστικά ομοιάζονται με τι αεροτρές εξάσει της ε, Εσθονίας. Επίσης, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ γειτονικέ του αγορέ οι οποίες δεν επιδοτούνται, από την άλλη αγορές οι ευρωπαϊκές εξακολουθούν και επιδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, φαντάζομαι ότι θέλουν να διαφοροποιήσουν απλώς την ε, οικονομία τους, ουσιαστικά να καταστήσουν ε, την οικονομία τους πιο ανταγωνιστική, να έχουν παρουσία σε περισσότερες περιοχές του κόσμου. Ακούσαμε επίσης και τη συμφωνία αυτή που υπήρχε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Νέας Ζηλανδίας πριν την προσχώρηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τελικά συμφωνία δεν είχε θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό το λόγο τελικά καταργήθηκε. Καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο οι δύο αυτέ χώρε, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, όσον αφορά το ζήτημα τη εποχικότητα. Για παράδειγμα, τα ακτινίδια. Ξέρω ότι υπάρχουν Ιταλοί και Γάλλοι παραγωγοί ακτινιδίων, οι οποίοι επενδύουν πάρα πολύ στη Νέα Ζηλανδία και θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό τον παράγοντα της εποχικότητας. Δεν πειλεί εμπορικό φραγμό αναγκαστικά. Και όσον αφορά την ε, ρυθμιστική ε, προστασία. Όσον αφορά λοιπόν τα πρότυπα, τα ρυθμιστικά πρότυπα και τα πρότυπα τα οποία διέπουν τα βασικά προϊόντα που έχουμε από τις οικονομίες αυτές. Βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί πάλι μία απόκληση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Άρα η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία ουσιαστικά δεσμεύονται από τη δική τους ε, ενιαία αγορά, από τις ε, περιφερειακές ε, συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Άρα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Και όσον αφορά τις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νομίζω ότι εδώ πέρα και ιδίω πριν τα Χριστούγεννα θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι πόροι που δίνονται για την επεξεργασία των δύο αυτών συμφωνιών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σας. Ο κύριος Πέζονεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανεξάρτητα με την δομή υποστήριξη του γεωργικού τομέα που υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο οι γεωργοί καλούνται να έχουν μεγαλύτερα κέρδη άμεσα από τους ίδιους τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές κατά κάποιο τρόπο έρχονται να αντικαταστήσουν τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν όλο και περισσότερους ενδιασμούς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό της υποστήριξης του γεωργικού τομέα, ιδίως στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Όταν ε, μιλάμε για τη γενικότερη εικόνα του ε, εμπορικού κλάδου που έθιξαν και ορισμένοι συνάδελφοι από την Επιτροπή, θα ήθελα προς αυτό να πω ότι ε, οι συνεταιρισμοί των γεωργών υποστηρίζονται πολύ συχνά από διάφορες πολυμερείς συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕΛΑ και στα πλαίσια διμερών συμφωνιών. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι τα πάντα θα ευθυγραμμίζονται, ότι θα υπάρχουν κοινά πρότυπα και κοινοί κανόνες και νομίζω ότι αυτό άλλωστε θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. Αυτό μας απασχολεί όλους ιδιαίτερος. Από την άλλη ακούσαμε και κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τη σύντομη δική μου παρουσίαση όσον αφορά την εποχικότητα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Μπορούμε να προσεγγίσουμε λίγο πιο στενά το ζήτημα. Το πρόβιο κρέας, για παράδειγμα, επηρεάζεται από την εποχικότητα. Πολλές φορές είχε θετικές επιπτώσεις το ζήτημα αυτό. Για παράδειγμα υπάρχουν περίοδοι όπου καταναλώνεται πολύ πρόβιο κρέας στην Ευρώπη. Και η όλη αυτή τάση έχει αντισταθμιστεί από περιόδους κατά τις οποίες δεν έχουμε ιδιαίτερα υψηλή πώληση τέτοιων προϊόντων. Και βέβαια αυτό επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Έχουμε κάποιες εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία ή την Αυστραλία που έχουν ε, ταράξει την ευρωπαϊκή αγορά πρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βέβαια έχει επηρεάσει αρνητικά πολλούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους μάλλον, οι οποίοι παράγουν κυρίως πρόβειο κρέας και εξαρτώνται ουσιαστικά από αυτό. Βέβαια για τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν καταναλώνουν πολύ πρόβειο κρέας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαμε δει ότι πολλές φορές ε, οι ε, εμπορικές τάσεις ε, που υπάρχουν παγκοσμίως επηρεάζονται από την ίδια τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Και ξέρετε ότι για παράδειγμα σε ορισμένε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά πρόβειου κρέατος έχει επηρεαστεί από αποφάσεις που ελήφθησαν στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από πολλούς συνεταιρισμούς εμπόρων. Δεν λέω ότι ευθύνουν αναγκαστικά οι εισαγωγές κρέατος από την Νέα Ζηλανδία ή την Αυστραλία. Ένα ακόμα στοιχείο, όσον αφορά το γάλα τώρα. Όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο αυτό. Η Φοντέρα είναι παρούσα στην Ευρώπη, επενδύει σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν μια κοινή δράση όσον αφορά τον τομέα αυτό. Αν δούμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε πώς αυτά θα επηρεάσουν τη στάση που θα κρατήσουμε στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Η παραγωγή γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή. Παράγουμε μεγάλες ποσότητες νοπού γάλακτος που διανέμεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διανομείς μας και βέβαια τα πράγματα δεν ακολουθούν αυτό το δρόμο στη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει μια άλλη διάρθρωση, προωθούνται άλλα προϊόντα όπως το αποκορυφωμένο γάλα και μιλάμε και διαφορετικές ποσότητες. Νομίζω ότι στη Νέα Ζηλανδία έχουμε 10 με 12 εκατομμύρια τόνους σε τήσια βάση όσον αφορά τον οπό γάλα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 116 εκατομμύρια, μάλλον 160 εκατομμύρια τόνους. που ουσιαστικά δεν ε, κινδυνεύουν, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα επηρεαστούν από μια νέα συμφωνία που θα έχουμε με τη Νέα Ζηλανδία. Πολύ φοβάμαι ότι ήδη η επικείμενη αυτή συμφωνία έχει αρχίσει να ασκεί πίεση στους Ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς. Και ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια ολόκληρη αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό μήνυμα λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά το γαλακτοκομικό τομέα και το πρόβιο κρέας και θα πρέπει να γνωρίζουμε τελικά πώς η νέα αυτή συμφωνία ενδεχομένως να επηρεάσει το επίπεδο τιμών στους κλάδους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα περάσουμε στην Αυστραλία και θα ήθελα αμέσως να δώσω το λόγο στον Justin Brown, τον απληρωτή γραμματέα εμπορίου από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω σήμερα στην Επιτροπή σας. Η κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού την Αυστραλία, της Αυστραλίας και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου τονίζουν τις ε, θερμές σχέσεις Αυστραλία και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεσμευόμαστε να εργαστούμε με την ε, Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για μια σύντομη έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και ε, ελπίζουμε στην συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία αυτή θα προωθήσει ένα ισχυρότερο εμπόριο στα αγαθά και στις υπηρεσίες, αλλά και ένα, μια αμφίδρομη εμπορική και επενδυτική σχέση και επίσης θα παίξει ένα ρόλο στην ενίσχυση της συνεργασίας ε, όπως την ε, νομοθεσία, την ψηφιακή οικονομία, την έρευνα, την ε, καινοτομία και άλλου. Σε Μια τέτοια συμφωνία επίσης θα τονίσει το γεγονός ότι η Αυστραλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη συνεργάζονται για πάρα, πολλά, ε, για πάρα πολλές στοιχείες του διεθνούς εμπορίου. Έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον στη στήριξη ενός ε, πολυμερούς εμπορικού συστήματος με ισχυρούς κανόνες που θα συμπεριλαμβάνουν και τον ΕΠΟΕ. Επίσης συνεργαζόμαστε για να προωθήσουμε διάφορες πρωτοβουλίες ε, συμπεριλαμβανομένης της ε, ε, συμφωνίας για τις υπηρεσίες και τα περιβαλλοντικά αγαθά αλλά και της ε, συμφωνίας για την, ε, για την ε, τεχνολογία των, της πληροφορικής. Επίσης, προσπαθούμε να προωθήσουμε την οικονομική ολοκλήρωση στον χώρο Ασίας Ειρηνικού και να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ολοκληρώσει τις διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα και είμαστε μία από τις 12 χώρες που ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο για την συμφωνία TPP. Ε, στο μέλλον επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με την Ινδία για μία διμερή ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης και συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία RCEP που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Και στις αρχές του επόμενου έτους θα συνεχίσουμε τις διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία. Η Αυστραλία λοιπόν έχει ε, μια πάρα πολύ ισχυρή υποδομή έτσι ώστε να στηρίξει και να προωθήσει την ανάπτυξη στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την, ε, της τεχνολογική, την τεχνολογική διασύνδεση στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ε, προσπαθούμε να χτίσουμε και για να κάνουμε ακόμα πιο ισχυρούς ε, τους δεσμούς που ήδη υπάρχουν. Είμαστε η έβδομη μεγαλύτερη αγορά στις υπηρεσίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι ένας ε, πολύ ελκυστικός προορισμός για τις επενδύσεις από την Αυστραλία και είναι η μεγαλύτερη ε, πηγή ε, επενδύσεων από το εξωτερικό. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιθυμούν η Αυστραλία να γίνει μια νέα βάση, ένα εφαλτήριο για να συνδέσει τα εμπορικά δίκτυα στην περιοχή μας. Ο στόχος μας ε, στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι να δημιουργήσουμε μια συμφωνία υψηλής ποιότητας που θα δώσει ένα, ε, μια περιεκτική ε, συμφωνία και ένα πολύ γόνιμο επενδυτικό περιβάλλον. Βλέπουμε επίσης πως είναι πάρα πολύ σημαντική η κατάργηση των εθελονιακών εδασμών και οι ε, διακρίσεις που δημιουργούν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις άλλες ε, χώρες. Οι δασμοί στην Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά χαμηλοί κατά μέσο όρο. Υπάρχουν όμως ορισμένοι τομείς όπου επιμένουν οι υψηλοί δασμοί. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ε, μια διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ίσο και δίκαιο εμπόριο στα τρόφιμα και στα γεωργικά προϊόντα το 2014 οι εξαγωγές της Ένωσης σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα στην Αυστραλία ε, ανέρχονταν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ε, αντίστροφα οι εξαγωγές της Αυστραλίας ε, ανέρχονταν περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς ανυπομονούμε να, ανοίξουμε, να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τα γεωργικά προϊόντα και σχετικά με τις υπηρεσίες η Αυστραλία επίσης ε, αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα απελευθερώσει ε, τις υπηρεσίες και θα άρει τους φραγμούς σε, ε, πολλούς, σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Η προτίμησή μας είναι η αναλήψη υποχρεώσεων να καταγράφονται σε, μια, σε έναν αρνητικό ε, κατάλογο και να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα προωθεί την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των αδειών σχετικά με τις επενδύσεις. Η Αυστραλία έχει μια μακρά ιστορία ε, θετικής αντιμετώπισης στο ξένο κεφάλαιο, στις ξένες επενδύσεις και επιθυμούμε ένα αποτέλεσμα, μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα ε, παρέχει διατάξεις που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και θα παρέχουν τις, ε, την κατάλληλη προστασία και ασφάλεια για τους επενδυτές και ταυτόχρονα θα προστατεύουν την ικανότητα της κυβέρνησης ε, να ε, λειτουργεί ως αριθμιστικός παράγοντας προς το κοινό συμφέρον. Επίσης, σχετικά με το ISDS, η κυβέρνησή μας θεωρεί πως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά, ε, και να εξετάζονται κατά περίπτωση. Έχουμε συμφωνήσει να συμπεριλάβουμε το ISDS στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που θα διαπραγματευτούμε και θα καλύπτουμε ορισμένους τομείς όπως ε, ε, η υγεία, το περιβάλλον και η, κρατική, η δημόσια πολιτική. Επίσης, θέλουμε να δοθεί έμφαση στην προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερης γραφειοκρατίας. Η, Αυστρία και η Αυστραλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια κοινή και πολύ ισχυρή πλατφόρμα υφιστάμενων ε, μηχανισμών και μέσων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το νομοθετικό μας ε, έργο στη συμφωνία αυτή. Ε, έχουμε ισχυρούς, ισχυρές βάσεις για το εμπόριο αλλά και για την ε, βιοασφάλεια και την ε, ασφάλεια των τροφίμων. Και επίσης συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της ανάπτυξης διεθνών προτύπων μέσω των Διεθνών Οργανισμών Δημιουργίας Προτύπων. Είμαστε επίσης ενεργό μέλος του ΠΟΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Πραγματικής Ιδιοκτησίας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε δεσμευμένοι για τη δημιουργία ενός πολυμερού συστήματος πολυ... πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα ε, κάτω από την συμφωνία TRIPS. Η δική μας προσέγγιση είναι να υπάρχει μια ισορροπία που θα χρησιμοποιεί ε, όλα τα δυνατά μέσα για το συμφέρον όλων. Επίσης, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση σε ορισμένα κεφάλαια που αφορούν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστήματων, ε, συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, όσον αφορά την γεωγραφική, ε, τις γεωγραφικές ενδείξεις, καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον χώρο και σκοπεύουμε να ε, σεβαστούμε τις επιθυμίες αυτές. Στην Αυστραλία υπάρχουν ορισμένες, ε, ορισμένα προϊόντα γεωγραφικής, ε, με γεωγραφικές ενδείξεις όπως το προσούτο, τα τυριά ροκφόρ, παρμεζάνα κτλ. Επίσης να σας πω ότι ιστορικά έχουμε έναν κοινό, ε, κοινή ιστορία και πρέπει να έχουμε και στο μέλλον έναν κοινό στόχο, τη δημιουργία δηλαδή μιας περιεκτικής και φιλόδοξης συμφωνίας σχετικά με τις ε, δημόσιες προμήθειες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για να προσχωρήσουμε στην ε, ε, Παγκόσμια Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες και ε, Επίσης, να σας πω ότι οι πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είχαν καλύψει και το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο στόχος μας, ε, πιστεύω, ο στόχος μας πιστεύω και η προσέγγιση μας είναι κοινή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι οι συμφωνίες είναι κάτι το περίπλοκο και είναι αναπόφευκτο και οι δύο πλευρές να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που θα αφορούν ευαίσθητα ζητήματα για τον κάθε φορέα και θα υπάρχει και αντίδραση από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Γι' αυτό λοιπόν ε, ελπίζουμε στην ε, ε, ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να καταλάβει ο καθένας την άλλη πλευρά όσο το δυνατόν περισσότερο. Πιστεύουμε στην Αυστραλία πως η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμφωνία που έρχεται σε την κατάλληλη στιγμή και θα ωφελήσει το παγκόσμιο, τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα χαρούμε πολύ για, ε, σε, να συνεργαστούμε στο μέλλον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάρ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σε αυτή την πρώτη φάση θα περιορίσω τις παρατηρήσεις μου σε κάποια γενικά θέματα και θα προσπαθήσουμε να δούμε το τι μας περιμένει μέχρι τώρα βλέποντας το τι έχει γίνει μέχρι τώρα όχι μόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε σχέση με το TPP. Εμείς είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους μας στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πω ότι ούτε εμείς ούτε ε, αυτοί δεν θα θέλαμε να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση όπως το TPP έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία αντιμετώπιση του θέματος η οποία ε, συνοψίζεται στη φράση «εμπόριο για όλους», «trade for all». Εμείς θα θέλαμε όμως αυτό να δούμε να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν μία θέση στους θεσμικούς μηχανισμούς ή συμφωνίας. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για διαφάνεια στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια πολύ θετικά βήματα σε σχέση με το TTIP και θα θέλαμε μια αντίστοιχη ε, προσπάθεια δεκτικότητας να διευρυνθεί και στις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ε, και επίσης και με άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία. Ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προτάσεις πρώτη για τα θέματα των ρητρών ή των κεφαλαίων ακόμα αηφόρου ανάπτυξης σε αυτές τις συμφωνίες. Σε σχέση με, με τον χώρο της εργασίας βασικό κλειδί θα έλεγα είναι η επικύρωση και πλήρης ε, και συνολική εφαρμογή ε, των συμβάσεων του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, σε σχέση επίσης και με τον ελάχιστη αμοιβή όπως επίσης και, τον ελάχι, και την ελάχιστη αμοιβή. Ε, δεν έχουν ε, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επικυρώσει την Σύμβαση 138. Δεν έχουν επικυρώσει επίσης και την 37. οι τροπολογίες σε αυτές τις νομικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν να αποκλίνουμε από τις βασικές αρχές του ILO. E του ILO. Ε, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λέγαμε ότι σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη συμπερίληψη των κεφαλαίων για την αηφόρο ανάπτυξη δεν έχουν γίνει πλήρες αντικείμενο εξετάλευσης ακόμα. Επίσης δεν έχουμε δει τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα σε χώρες όπως η Κορέα που ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ή και σε άλλες χώρες όπως η Γουατεμάλα και η Σουαζιλάνδη. Όπως και να έχουν τα πράγματα η απουσία οικονομικών συνεπειών για τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων ε, θα έλεγα καταδικάζει την πρόταση αυτή σε ένα επίπεδο καλών προθέσεων. Θέλουμε εμείς να καλύψουμε όλους, ε, όλες τις πιθανές ε, παραβάσεις και ε, παραλήψεις σε, στα εδάφη όλων των συμμετεχόντων. Θα πρέπει να συνδέονται επίσης οι ευθύνες των επενδυτών με την προστασία των επενδυτών όπως ο κώδικας του ΟΣΑ ε, για τις ε, πολυμερείς ε, συμφωνίες, όπως επίσης και οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την επιχειρηματικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πρότασή της για το TTIP η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι το σύστημα CSR είναι εθελοντικό, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει και έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από πλευράς της Νέας Ζηλανδία ε, και ε, της Αυστραλίας ε, δεν δείχνουν παρά το ότι πράγματι οι χώρες αυτές είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με διαφορετικό τρόπο αλλάζοντας τις προηγούμενες θέσεις τους. Όπως γνωρίζουν τα μέλη της ΣΥΝΤΑ, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι κατά ε, των ε, ρυθμίσεων του ISTS, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν διευκολύνει, ε, επιβάλλει μάλλον κάποια μέτρα εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εθνικών αμυγός επιχειρήσεων και όχι στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το νέο σύστημα SCS εξακολουθεί να κάνει την διάκριση ανάμεσα ε, σε τοπικούς και ε, σε τοπικούς επιχειρηματίες και ξένους επιχειρηματίες. Υπάρχουν θέματα ε, όπως αυτά τα οποία καλύπτουν την παραγωγή καπνού και νομίζω ότι κάθε πρόκληση για συλλογικές συμβάσεις που να εξαιρούνται είναι απαράδεκτες και δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη στα κοινωνικά θέματα και να πληρώνει τους φόρους της. Σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, να διατηρηθεί η ισχύουσα πρακτική και να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες ο σεμβασμός της Σύμβασης 84 του ILO για τις, δημόσι... για τις συλλογικές συμβάσεις σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες πρέπει να είναι η αναφορά για όλες τις συμφωνίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της παραγής φαρμάκων με χαμηλό κόστος, της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν θα πρέπει να υπονομευθούν μέσω του ανοίγματο της αγοράς. Οι ρυθμίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις συλλογικέ μας προτιμήσεις. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Δεν είναι έτσι όμως, όπως και δεν, είναι, ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και για την απελευθέρωση των αγορών. Όπως ε, ε, προτείνουμε εμείς, ε, ε, δεν θέλουμε να καταργηθούν πλήρως όλες οι μορφές εμποδίων, αλλά θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ευθυγράμμιση στα επίπεδα προστασίας θα πρέπει να είναι προς τα πάνω. Και δεν μπορεί να υπάρξει ε, και πρέπει μάλλον να μπορεί να υπάρξει μια ρήτρα που να απαγορεύει την παραβίαση αυτών των κανόνων. Θα πρέπει να εμπλακούν επίσης οι κοινωνικοί εταίροι και στις συζητήσεις για τους θεσμικούς αυτούς μηχανισμούς. Το, η Συνομοσπονδία λοιπόν των Συνδικάτων επιθυμεί και επιμένει να εμπλακεί σε ανοιχτές συζητήσεις ε, με όλους τους υπόλοιπους εταίρους. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε τον χρόνο σας. Ο Πασκάλ είναι τελευταίος ομιλητής από το European Services Forum. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Πρέσβης, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Να σας πω ότι δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για την Γεωργία και η συμφωνία αυτή πιστεύω τελικά θα έχει να κάνει κυρίως με τις υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 1,73% το έπτης ε, που καλύπτεται από υπηρεσίες, 67,4% για την Αυστραλία, 69,6% για τη Νέα Ζηλανδία. Οι υπηρεσίες λοιπόν αυτές αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα των συμφωνιών αυτών. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό εμπόριο υπηρεσιών. Έχουμε πάνω από 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που αποτελούν πλεόνασμα του ευρωπαϊκού εμπορίου στις υπηρεσίες. Πολύ σημαντικά ποσά αυτά σε σχέση με τα όσα ακούσαμε για τη Γεωργία. Επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι εξαγωγές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αζηλανδία και την Αυστραλία είναι πολύ ψηλές. 41% του συνολικού εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας αντιστοιχεί σε υπηρεσίες. Για τη Νέα Ζηλανδία το ποσοστό αυτό είναι 32% και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Επίσης, οι επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη επενδύει άμεσα πολύ σημαντικά στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία με 122 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Και νομίζω ότι θα θέλαμε να δούμε και περισσότερες επενδύσεις αμφίδρομες, δηλαδή από την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Όσον αφορά τώρα την απασχόληση, μολονότι οι υπηρεσίες όπως είπα αντιστοιχούν στο 69% του ΑΕΠ της Αυστραλίας, στο 83% των θέσεων απασχόλησης στην Αυστραλία και στην Ζηλανδία, ένα αντίστοιχο ποσοστό είναι θέσεις απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και η δική μου οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υπηρεσιών, θέλει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό αυτές τις διαπραγματεύσεις, αρκεί για να διορθώσουμε κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Προκαλεί εντύπωση το γεγονό ότι η Αυστραλία, και η Νέα Ζηλανδία δεν έχουν συνάψει διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε με πολλέ άλλε χώρε. Ένα από τα επιχειρήματα που ακούσαμε είναι ότι οι δύο αυτέ χώρε ουσιαστικά έχουν την ίδια νοοτροπία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκουν στον ΩΣΑ, ακολουθούν του ίδιου κανόνε με αυτού που ισχύουν στον ΩΣΑ, συμμετέχουν στι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Τίζα, όπω ακούσαμε πριν από λίγο. Είναι δύο χώρε οι οποίε ε, θα συνάψουν επίσης και τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Έγινε μια νέα προσφορά από την Αυστραλία. Ήδη η Νέα Συλλανδία έχει συνταχθεί στη συμφωνία αυτή ήδη από πέρυσι. Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας δύο χώρες που έχουν μια κοινή νοοτροπία με αυτή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Στην πράξη λοιπόν ο οργανισμός μου, το ESF, υποστηρίζει τις δύο αυτές συμφωνίες και λέμε μάλιστα ότι θα πρέπει να έχουμε και σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Δηλαδή θέλουμε ουσιαστικά ένα ενισχυμένο GATS, GATS+. Plus. Η βάση των δύο αυτών συμφωνιών θα είναι καταρχάς οι δεσμεύσεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας όσον αφορά τον GATS. Είναι μέρη της ΤΙΖ επίσης οι δύο αυτές χώρες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μια συμφωνία η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια βελτιωμένη μορφή της τίζα, τίζα πλάσα. Εφόσον όμως η τίζα θέλει να πάρει τη μορφή της καλύτερης δυνατής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, θα πρέπει να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία που θα είναι TPP+, ουσιαστικά μια βελτιωμένη μορφή της συμφωνίας εμπορικών σχέσεων στο χώρο του ειρηνικού. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει η συμφωνία αυτή να αποτελεί και GPA+. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να προσχωρήσουν στο GPA, στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά όπως και με τον Καναδά θα θέλουμε είτε να μειώσουμε το κατόφλι. Ξέρετε ότι ε, στην ε, Ευρώπη δεν μιλάμε για κυβερνητικές συμβάσεις αλλά για δημόσιες συμβάσεις. Ουσιαστικά αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε, όλες τις, σε όλους τους δημόσιους φορείς και όχι μόνο στους κυβερνητικούς φορείς. Ξέρετε ότι ε, σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές υπηρεσίες τις οποίες θέλουμε να εντάξουμε στη συμφωνία αυτή. Τι μορφή θα πρέπει να πάρουν τώρα διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργό Εμπορίου. Θέλουμε και εμείς να έχουμε αρνητικό κατάλογο. Είναι δύο αναπτυγμένες χώρες, η Νέα Ζηλανδία και, ο... και η Αυστραλία. Θέλουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ακολουθούμε και με τον Καναδά και με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Πλήρη δηλαδή αρνητικό κατάλογο. Στην πράξη θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως την κατάσταση, να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή μορφή FTA ή GATS ή να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Να έχουμε δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά το εφιστάμενο ρυθμιστικό επίπεδο. Σε άλλους τομείς θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ευέλικτους κανονισμούς. Σας δώσω κάποια παραδείγματα προς τα που θέλουμε να κινηθούμε. Σε οριζόντιο επίπεδο, όταν διαπραγματευόμαστε για τον τομέα των υπηρεσιών, μιλάμε για διασυνοριακές υπηρεσίες. Και ξέρετε ότι βέβαια έχουμε εδώ το περίφημο, την περίφημη διασυνοριακή ροή δεδομένων. Η δική σας επιτροπή κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπόριο χωρίς την διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων. Τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου πλέον χωρίς να υπάρχουν δύο υπολογιστέ που θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Θέλουμε λοιπόν οι εμπορικέ αυτέ συμφωνίε να διασφαλίζουν ότι όντω θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε διασυνοριακή ροή δεδομένων συγκεκριμένους κανόνες όπου δεν θα έχουμε υποχρέωση εγκατάσταση σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένου κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της συμφωνίας αυτής. Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα στις εμπορικές αυτές συμφωνίες που έχουν να κάνουν κυρίως με τον κλάδο υπηρεσιών και που επηρεάζουν τελικά οποιοδήποτε κλάδο, γεωργικά προϊόντα, ή άλλους τομείς όπως η μεταποίηση είναι η προσωρινή κινητικότητα των εργαζομένων, η προσωρινή κινητικότητα των παρόχων υπηρεσιών αλλά και προσωρινή κινητικότητα μηχανικών για παράδειγμα που πηγαίνουν από τον τόπο μεταποίησης προς τον πελάτη, εκεί δηλαδή όπου παρέχονται συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Με την Αυστραλία λοιπόν και τη Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μία συμφωνία η οποία θα μας επιτρέπει να προασπίσουμε τους τομείς αυτούς, να προωθήσουμε τον τομέα των υπηρεσιών και να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση αδειών, προσόντων και δεξιοτήτων. Κατά αυτόν τον τρόπο δικηγόροι, αρχιτέκτονες ή ελεγκτές μηχανικοί θα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν προς τις χώρες αυτές και αυτόματα να γνωρίζονται τα προσόντα τους. Αυτό θα αποτελέσει σαφώς προστιθέμενη αξία αυτής της συμφωνίας. Τώρα όσον αφορά τους διάφορους τομείς. Προφανώς θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο τι έχουμε πετύχει στα πλαίσια της TPP, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι ταχυμεταφορές, οι υπηρεσίες ε, διανομής προϊόντων, επαγγελματικές υπηρεσίες όπως οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ε, λογιστών, ελεγκτών, η, η Αυστραλία, με συγχωρείτε, ενδιαφέρεται επίση για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, ιδίω για τον τομέα τη λιανική τραπεζική, καθώ επίση και τον τομέα, τον τομέα των ασφαλίσεων. Στα πλαίσια της ε, TPP δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ δεσμεύσει όσον αφορά την αεροναυπηγική, τις θαλάσσιες μεταφορέ. Εμεί όμω θα μπορούσαμε να καλύψουμε και αυτού του τομεί στη συμφωνία μα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντα, να πω κάτι που είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε συγκεκριμένο κεφάλαιο όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Το έχουμε πει αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει σε κάποια κεφάλαια να έχουμε μία μείωση της προστασίας των επενδύσεων και όσον αφορά την συνεργασία στον ρυθμιστικό τομέα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε δοκιμάσει με την Αμερική και νομίζω ότι και με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να έχουμε μια κοινή διαδικασία όσον αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τρεις συναδελφούς που ζήτησαν το λέγω. Ο κύριος Κέλνερ πρώτος. Ευχαριστώ. Άκουσαμε με μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί είναι καλές οι διατάξεις ε, της TTP ε, για την προστασία των ε, επενδύσεων. Τις διάβασα. Και αυτή είναι μία ερώτηση που αφορά ένα ευαίσθητο θέμα για την Αυστραλία. Γιατί λοιπόν αυτές οι ε, διατάξεις είναι καλές από τη δική σας ε, ε, οπτική γωνία. Επίσης, για το e θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σας απασχολεί η επικύρωση όπως μας είπατε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της ελευθερίας, ε, του δικαιώματος του συνέχεσθε είναι θέμα αρχής. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα του κατώτατου μισθού. Και επίσης, ε, μας είπατε αυτά που δεν θέλετε, αλλά θα ήταν περισσότερο ενδιαφέρον να μάθουμε τι είναι αυτά που θέλετε. Ακούσαμε για την διοργάνωση και τα λοιπά, αλλά τα μέλη αυτών των οργανισμών χρειάζονται δουλειές και γι' αυτό λοιπόν αυτές οι δουλειές, αυτές οι θέσεις απασχόλησης πρέπει να δημιουργηθούν. Είναι πιστεύω γενικότερο το συμφέρον αυτό. Έπειτα μας είπατε ότι σας απασχολεί η εναρμόνιση και θυμάμαι και όλα σε αυτό που είπατε, ότι η γραφειοκρατία, ότι για κάποιους είναι γραφειοκρατία, για κάποιους είναι κόκκινη γραμμή. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτές οι συζητήσεις σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας κτλ. Μπορείτε να μου πείτε ε, κατά τη δική σας ε, άποψη πώς εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν αυτές ε, οι χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όντω πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Αυστραλία, διότι ο γιος μου είναι εκεί και έχουμε λοιπόν πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλές στενές σχέσεις με τη χώρα. Τώρα σε σχέση με τις εμπορικές ε, συμφωνίες που συζητάμε, είναι πιθανόν, είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία με την Αυστραλία και όχι με την Νέα Ζηλανδία ή το αντίστροφο. Και ποιες θα ήταν οι συνέπειες για κάθε μία από αυτές τις χώρες που θα είναι εκτός συμφωνίας. Επίσης, ε, η κυρία Καρ αναφέρθηκε σε κάποιες προτάσεις της κυρίας Μάλιμστρομ. Όμως είπατε ότι παραμένουν κάποιες δυσκολίες για τις εγχώριες επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν για τις ε, πολυεθνικές, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Και τέλος, σχετικά με τη ροή δεδομένων. μήπως υπάρχει φόβος ότι στην Ευρώπη είμαστε πολύ περιοριστικοί σχετικά με τις ερωές ε, δεδομένων και πώς ε, περιορίζουμε τα πράγματα παρά τα απελευθερώνουμε. Ε, ο David Martin. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα είμαι σύντομος η ομάδα μου συμφωνεί απόλυτα. Χρειαζό, χρειάζεται ένα κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης και για τις δύο συμφωνίες, αλλά για όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει ένα ε, κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ο κύριος Πασκάλ είχε απόλυτο δίκιο. Οι υπηρεσίε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, συμφωνίας και αναφερθήκατε και σε αυτόν τον αρνητικό κατάλογο και εγώ πιστεύω πως καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ένα θετικός κατάλογος. Το πιστεύω εγώ, το πιστεύει και η ομάδα μου. Ε, επίσης, θα ήθελα να μάθω εάν πιστεύετε πως θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ε, κάτι επιπλέον, κάποια επιπλέον συμφωνία που δεν μπορούμε να καλύψουμε με την συμφωνία ΤΙΣΑ. Γιατί λοιπόν θεωρείτε πως μια διμερή συμφωνία είναι πιο σημαντική από τη συμφωνία ΤΙΣΑ. Και τέλος, όπως ρώτησαν και άλλοι, έχει να κάνει με, με το ISDS. Φυσικά δεν διαπραγματευόμαστε εδώ, αλλά θα ήθελα να μάθω την άποψή σας και αν το ISDS μπορεί να ενταχθεί στο υφιστάμενο μοντέλο που υπάρχει στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή. Ο Ντάνιελ. Έχω μία ερώτηση για την ε, κυρία Κάρ. Αναφέρθηκε στη διαφάνεια. Θα ήθελα ο κύριος Κένας και η κυρία Κάρ να μου απαντήσουν στο εξής. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο διαδίκτυο διάφορα έγγραφα διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP. Εσείς, μετά από αυτό, έχετε κάποιο παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσφέρει διάφορα τα οποία είχε αρνηθεί δημόσια. Μπορούμε σε αυτά τα έγγραφα δηλαδή να βρούμε κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις διαπραγματεύσεις και τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να τα προσφέρει. Θα ήθελα δηλαδή να επαληθεύσω με άλλα λόγια το, το τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντάρκμαουθ έχει το λόγο. Ναι, και εγώ, ε, και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα γιατί η γυναίκα μου ήταν από την Αυστραλία. Θα ήθελα και εγώ να εκδηλώσω ένα αντίθετο ενδιαφέρον, διότι η γυναίκα αυτή είναι, δεν είναι πλέον γυναίκα μου. Εκτιμώ το γεγονό ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ...μέσα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ στην οικονομία του. Αλλά δεν είναι σαφέ για μένα το εάν πρέπει να συνδυαστούν αυτές οι δύο συμφωνίες, να συνδεθούν. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε να είναι ξεχωριστές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε περισσότερα γι' αυτό. Και οι υπόλοιπε ερωτήσει μου είναι παρόμοιε με τις προηγούμενες. Ε, Δυστυχώ δεν προλάβατε να ε, τις ε, αναπτύξετε. Αναφέρομαι στα τρία σημαντικά στις τρεις σημαντικές ε, χώρες, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, που δεν έχουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι λοιπόν αν είναι απαραίτητες αυτές οι συμφωνίες. Χρειάζονται αυτές οι συμφωνίες. Ε, δεν θέλω να σας ε, εκθέσω ή να σας φέρω σε δύσκολη θέση, όμως θα ήθελα να μου απαντήσετε. Και έπειτα θα με ενδιέφερε να μάθω ποιες θα θεωρείτε πως είναι οι ε, θετικές ε, συνέπειες της Συμφωνίας Αυστραλίας-Κίνας. Και κάτι τελευταίο. Και ο κύριος Γκρόσερ και ο κύριος Πράν ε, έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι για να φτάσουν εδώ και μου φαίνεται κάπως περίεργο ε, το ότι η Επιτροπή αυτή έχει αφιερώσει τόσο λίγο χρόνο σε αυτούς τους καλεσμένους και τόσο πολύ χρόνο σε εκπροσώπους από λόμπι. Ο κύριος Τάκουλα. Άκουσα τους συναδέλφους, άκουσα και τον Ντάρθμουθ. Είναι κρίσιμη η εποχή για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που επιθυμούν εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εσείς ενδιαφέρεστε για να συνδεθούν οι χώρες αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσείς θέλετε να φύγετε η δική σας χώρα από την Ένωση, εν πάση περιπτώσει. Μια ερώτηση για τον κύριο Μπράουν. Ασχοληθήκατε και με τις διαπραγματεύσεις λοιπόν για το TTP. Ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το πιο βασικό επίτευγμα για το TTP και ποιος είναι πιστεύετε ο ρόλος της Αυστραλίας στις διαπραγματεύσεις αυτές λόγω μεγέθους. Σύντομα Πρόεδρε, ο κύριος Κάμπελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προσπαθήσει να επιβάλλει παλαιότερα στα θέματα της διαπραγμάτευσης τις απόψεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σε καμία περίπτωση ε, ανεκτό από πλευράς τους. Και τα ίδια προβλήματα έχουμε και με τη ΣΕΤΑ, ε, πάντα για το ίδιο θέμα των περίφημων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς μιλάμε για εμπόριο και για θέσεις απασχόλησης και όχι για πολιτική. Προφανώς πρέπει να θέσουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά να μην τα συγχαίρουμε. Και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των, των συνδικάτων μάλλον, έθεσαν τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων κτλ. Όχι, δεν είναι εδώ ο χώρος. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης και όχι να χάνουμε το χρόνο μας συζητώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέσσερα λεπτά κύριε Μπράουν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να δώσω όσο περισσότερες απαντήσεις μπορώ. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, γιατί εμείς υπογράψαμε στα πλαίσια του TPP τα θέματα της προστασίας, της ρήτες προστασίας των επενδυτών. Απλή είναι η απάντηση. Ήταν βασικό στοιχείο της συνολικής συμφωνίας και έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα δεχόμασταν αυτή την πρόταση ή να μην υπογράψουμε συνολικά τη συμφωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμπεριλήφθη και στο τελικό κεφάλαιο νομίζω και συνολικά ήταν κάτι το οποίο μπορούσαμε να δεχτούμε. η Επίτροπος Μάλστρομ ήταν ιδιαίτερα δεκτική σε σχέση με τα θέματα αυτά. Εμείς αναγνωρίσαμε κάποια από τα θετικά στοιχεία των προτάσεων τα οποία συμμεριζόμεθα. Η πολυδιάσπαση του συστήματος είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας και το οποίο θα συζητήσουμε και στο μέλλον. Και μια άλλη ερώτηση δεν ξέρω αν απευθύνεται σε μένα, αν θα έπρεπε δηλαδή να ληφθούν υπόψη οι προτιμησιακές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εμπορικούς της εταίρους. Ε, προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τέτοια συμφωνία με κάθε εμπορικό εταίρο μέσω του ΠΟΕ. Είναι πάντα ε, το πεδίο αναφοράς για τη συνεργασία ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους στα πλαίσια του ελευθέρου εμπορίου. Τώρα αν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω προτιμησιακού τύπου ιδιαίτερες συμφωνίες ανάμεσα σε εταίρους είναι κάτι το διαφορετικό. Τώρα για τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμφωνίας με την Κίνα. Μπορώ να σας δώσω στοιχεία για τις πιθανές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Ε, υπάρχουν από το TPP κάποια πολλά θετικά και κάποια αρνητικά. Ε, ένα από τα ωφέλη είναι οι νέες προσβάσεις ε, ή μάλλον οι προσβάσεις σε νέες αγορές για πάρα πολλά προϊόντα. Είναι μια περιφερειακή συμφωνία και μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο σύστημα ε, γεωγραφικών ενδείξεων σαν παράδειγμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια συνεκτικότητα στον τομέα των διακανονιστικό, κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο για τους εξαγωγούς μας. Ε, είχαμε επίσης ε, κάποιες πολύ δύσκολες συζητήσεις για το θέμα της προστασίας των ε, ε, εμπιστευτικών δεδομένων για τη φαρμακοβιομηχανία. Ήταν δύσκολες ε, οι διαπραγματεύσεις αυτές. Τελικά καταλήξαμε σε κάτι το οποίο νομίζω είναι σχετικά ικανοποιητικό. Και τέθηκε και μια τελευταία ερώτηση για το τι είναι το σημαντικό για μας με αυτή την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα θέματα είναι υπό εξέταση, δεν κρύβουμε τίποτα, δεν αποκλείουμε τίποτα και στόχος μας είναι να υπάρξει μια σωστή ισορροπία με αμοιβαία ωφέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Λίνα Κάρ. Ευχαριστώ πολύ. νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβω κάποια πράγματα. Δεν είμαστε κατά του εμπορίου ως συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θέλουμε ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού και κοινού κανόνες, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνίζονται τις άλλες επιχειρήσεις βάσει κοινών κανόνων. Όσον αφορά τη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ξέρετε ότι πρόκειται για τα ελάχιστα εργασιακά πρότυπα τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, οποιαδήποτε δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό της θα πρέπει να μπορεί και να επικυρώνει αυτές τις συμβάσεις και να τις εφαρμόζει στην πράξη. Τώρα, πώς έχει κατάσταση με το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε επιτόπου. Επ' αυτού νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω, δεν γνωρίζω πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, πώς έχει το σύστημα εκεί, αλλά οι συνάδελφοι, ιδίω από τη Νέα Ζηλανδία, μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβλήματα με το εργασιακό δίκαιο της χώρας, το οποίο προβλέπει προτιμησιακή μεταχείριση και κάποιες εξαιρέσεις σε σχέση με τη σύμβαση του ILO όσον αφορά τον τομέα του εμπορίου. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι να βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία της προστασίας των εργαζομένων και των εργασιακών συνθήκων και άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για άνηση μεταχείριση, γιατί βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χαίρουν τέτοιων εξαιρέσεων, αλλά οι εμπορικοί μας εταίροι έχουν τέτοιες εξαιρέσεις για τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θέλουν να δημιουργηθούν προφανώς θέσεις απασχόλησης, Ουδέποτε εμεί ταχθήκαμε κατά τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ενδιαφερόμαστε κι εμεί πάρα πολύ για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία, όσο και εσεί εδώ πέρα. Το θέμα πάντως είναι τι είδου θέσει απασχόληση θέλουμε, τι εργασίε δημιουργούμε, επισφαλεί μόνο θέσει απασχόληση με χαμηλέ κοινωνικέ διασφαλίσει οι οποίες δεν διέπονται από θετικές εργασιακές συνθήκες ή δημιουργούμε τελικά θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητος που απευθύνονται σε υψηλά εξειδικευμένους εργαζόμενους. Και ποτέ εμεί δεν είπαμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ευθυγράμμιση κάποιων κανόνων με τους εταίρους μας. Το αντίθετο, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας τώρα. Προσωπικά δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια έγγραφα μυστικά τα οποία δεν είδαμε. Δώσαμε πραγματικά όμως μία μάχη στο παρελθόν προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Το TTIP είναι το καλύτερο παράδειγμα αν θέλετε. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά κοινοποιούσε, γνωστοποιούσε τα διαπραγματευτικά έγγραφα, αλλά παράλληλα εμείς δεν είχαμε καμία απολύτως πρόσβαση στις διαπραγματευτικές τοποθετήσεις και στα σχετικά έγγραφα των ΗΠΑ. Χρειάστηκε να καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες για να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τη διαπραγματευτική στάση της Ιαπωνίας. Η, διαφάνεια, η διαφάνεια λοιπόν ισχύει από τη Φέντη για το TTIP, αλλά δεν διέπει τις υπόλοιπες συμφωνίες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στις μελλοντικές συμφωνίες θα πετύχουμε το ίδιο επίπεδο διαφάνειας με αυτό που έχουμε τώρα για τη συμφωνία TTIP. Και σας είπα άλλωστε ότι ε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιθυμούν ε, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αρκεί αυτές να είναι ποιοτικέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κερνάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, τώρα, γιατί ένας αρνητικός κατάλογος και όχι ένας θετικός. Καταρχάς, ο αρνητικός κατάλογος είναι κάτι που δίνει περισσότερη διαφάνεια. Βλέπουμε τι δεν πρέπει να γίνεται και μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί ο θετικός κατάλογος είναι κάτι που χρησιμοποιούμε όταν διαπραγματευόμαστε με αναπτυσσόμενες χώρες, ε, οι οποίες έχουν λιγότερες δυνατότητες να αναλάβουν υποχρεώσεις σε ορισμένους τομείς ή υποτομείς. Όμως δεν νομίζω πως ε, με, κάποιες, με τις αναπτύγμενες χώρες ε, μπορούμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αρνητικό κατάλογο και στι πολυεθνικέ εταιρείε ισχύουν τα ίδια. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Τώρα, σχετικά με την ΤΙΖΑ και τις εδημερείς συμφωνίες και τι μπορούμε να ε, καταφέρουμε με τις εδημερείς που δεν μπορούμε με την ΤΙΖΑ. Καταρχάς, δεν νομίζω πως θα καταφέρουμε περισσότερα με την συμφωνία ΤΙΖΑ που ε, δεν θα έχουμε με τη συμφωνία TPP. Η πρόσβαση στην αγορά θα είναι περιορισμένη και Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μπορούμε να επιλύσουμε με την συμφωνία ΤΙΣΑ και αυτό είναι καλό, θα υπάρχει μια σχετική πειθαρχία. Όμως αν θέλουμε να εμφαθύνουμε τη συνεργασία μας, οι διμερείς συμφωνίες είναι ε, κατάλληλες. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η ΤΙΣΑ δεν αναφέρει καθόλου τις δημόσιες προμήθειες. Σχετικά με τη διαφάνεια τώρα. Θα συμφωνήσω με τον διπλανό μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργήσε με διαφάνεια και δεν υπάρχουν πολλά έγγραφα που δεν έχουμε δει. Φυσικά θα θέλαμε να δούμε περισσότερα έγγραφα από την άλλη πλευρά των ε, διαπραγματεύσεων της ε, συμφωνίας TTIP. Και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η επιθυμία για διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή επίσης ε, μην ξεχνάτε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και κανείς δεν έχει ζητήσει να δει τίποτα. Η διαφάνεια λοιπόν πιστεύω πως ε, πρέπει να αφορά όλους ε, εξίσου και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία σίγουρα ενδιαφέρονται να δώσουν ε, διαφάνεια σχετικά με τη ροή δεδομένων. Ε, και το αν υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ περιοριστική. Μπορώ να σας πω από τη δική μας πλευρά πως ε, θα θέλαμε να αποφύγουμε να γίνει πολύ περιοριστική η Ευρωπαϊκή Ένωση με την προστασία δεδομένων κτλ. Γι' αυτό και έχουμε τοποθετηθεί όπως έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θέλουμε να μεταφερθούν αυτές οι ε, αυτές οι ανησυχίες, αυτά τα προβλήματα σε μια συμφωνία. Αυτό που προσπαθούμε να κοιτάξουμε είναι ότι έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ροές δεδομένων που μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο και καλή συνεργασία στις δύο χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει τώρα να συνεχίσουμε στα αγγλικά, διότι έχουμε ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ τους διερμηνείς και συνεχίζουμε στα, γερμα... στα αγγλικά